Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ε, συγγνώμη που καθυστερήσαμε λιγάκι. Ε, προσπάθησα να διευθετήσω μερικά ζητήματα για την αποστολή στην Κρήτη, η οποία είναι μεγαλύτερη σε σύνθεση από την αποστολή ε, από την ομάδα που θα πάει στο ΑΚΕ. Θα ήθελα να συνεχίσω λοιπόν, συνεχίζοντας με τις ανακοινώσεις του Προέδρου και τα αποτελέσματα της ε, συνεδρίασης των συντονιστών. Όσον αφορά τους εισηγητές και συντάκτες υπάρχει μια πρόταση για την τροπο, τροποποίηση του 2019 2009 κάθετος 19 για τις γνωμοδοτήσεις πρόταση για την άμεση οδηγία για τις χώρες σημαία και τις ευθύνες τους και την υλοποίηση ε, του κανονισμού 13-2009 του Συμβουλίου που καλύπτει τη συμφωνία μεταξύ εφοπλιστών, πλειοκτητών δηλαδή και την Ένωση ε, Ναυτικών, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Ναυτικών, Ναυτεργατών. Για την πρόταση κανονισμού ανακύκλωσης ε, πλοίων, ανακύκλωσης σκαφών. Δεν θα κάνουμε τίποτα και η απόφαση για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Hong Kong ε, για την ανακύκλωση και πάλι των σκαφών, πλοίων. Δεν θα κάνουμε τίποτα ουδεμία δρόση όσον αφορά τώρα την ε, μεταφορά οχημάτων οι οποία έχουν, τα οποία έχουν καταχωριστεί σε πολλαπλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Working document program. ουδεμία δράση ε, ε έξεση προόδου επίσης ουδεμία δράση όσον αφορά την ΕΟΚΕ ε, και την έκθεση για την ε, Βαλτική το θαλάσσιο χώρο της Βαλτικής ουδεμία δράση, κοινή πρόταση για την ενεργειακή κοινότητα, πρόταση δηλαδή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την ενεργειακή, στο Συμβούλιο των Υπουργών για την ενεργειακή κοινότητα ουδεμία δράση. Όσον αφορά τώρα τη Συμφωνία των ε, Προεδρών των Επιτροπών για την προθεσμία ε, χρηματοδότησης της ΆΣΑ ουδεμία δράση. Η απόφαση για το πρόγραμμα εργασίας 2013 είπαμε ότι η προτεραιότητα θα είναι η Ευρωπαϊκή Ουρανή και η, αγορα, η αγορά, ε, συνθήκες εργασίας και συνθήκες εργαζομένων, ε, ηλεκτρονική εργασία, ε, ναυτιλία, ναυτιλια, θαλάσσιος χώρος, ναυτιλίες, ναυσιπλοεία κλπ. Και ο κύριος, η έκθεση του κυρίου Μπάτσε για τα δικαιώματα των επιβατών θα ψηφιστεί μετά την, ε, ε, την καλοκαιρινή διακοπή. Το σύστημα κρατήσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και ο νομοθετικός διάλογος, εκεί οι συντονιστές συμφώνησαν να το βάλουν στην μερίσια διάταξη για την επόμενη συνεδρίαση. Αυτή είναι λοιπόν η Αυτές είναι οι αποφάσεις των συντονιστών. Ε, υπάρχει κανένα σχόλιο παρακαλώ, ερώτηση. Ωραία. Τότε ε, συμφωνούμε ε, στην έξεση αυτή των συντονιστών και την επαναπέμπουμε στους συντονιστές. Επόμενο θέμα είναι οι ψηφοφορίες. Έχετε τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας παρακαλώ. Να κάνουμε μία δοκιμή γιατί συνήθως ε, έχουμε έναν-δύο πλεονάζοντες ε, που ψηφίζουν. Έχετε όλες τις κάρτες σας, πολύ ωραία. Να κάνουμε λοιπόν το τεστ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρα της ψηφοφορίας. Φαίνεται ότι το ΕΛΚ έχει το σωστό αριθμό ψήφων, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι η έκθεση του κυρίου Ζήλε, πρόταση οδηγίας για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη. Τροπολογία 16. Η 15 έχει αποσυρθεί. 16 ως ε, προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ηλεκτρονικός. άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. Δεκτή. Έπεται τροπολογία 4 του εισηγητή υπέρ. Κατά. αποχές Εγκρίνεται. 17 ως προσθήκη. Στο άρθρο 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. <clears throat> τροπολογία 5. Είναι συμβατή. Την ψηφίσαμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 18. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να φτιάξει και το τσάι μου, λέει ο πρόεδρος. 21. Κυρία Στικάου, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22. Προσθήκη, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23. Προφορική, προφορική, ψηφοφορία, ε, Είσαστε όλοι εντάξει ευχαριστημένοι με αυτή την προφορική. Τότε ψηφίζουμε την 23. <clears throat> Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 7. Και πάλι προφορική τροποποίηση, τροπολογία, εξαρισμός ε, θα παράσχεται κτλ. κτλ για να μην συσσωρεύονται τα εκρηκτικά αέρια. Ωραία. Ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ή 7 ήταν αυτή. Μπορεί κάποιος, ε, παρακαλώ, να μου φέρει νερό και γάλα για το τσάι μου. Εγώ φέρνω το φακελάκι του τσαγίου από το σπίτι μου, αλλά το νερό πέρασε μπροστά μου και δεν πρόλαβα. Ναι, ναι, 24 της κυρίας Ζαντόνκα, 24 παρακαλώ, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25, άχι διαγραφή, για διαγραφή, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 ο κ. Μασίνκεβιτς. Προφορική τροπολογία. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε την 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε παρακαλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος της τροπολογίας 9 με την προφορική ε, τροπολογία. Προφορική... Ψηφίσατε. έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 10. Και πάλι προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα. Υπάρχουν αντιρρήσεις στις προφορικές αυτές τροπολογίες, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 10, το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επιτέλους έχω το γάλα μου. Το, ε, το 15 η, 11 ή 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κάτι τρέχει με το γάλα. Η προμήθεια γάλακτος σήμερα πάσχει. Τροπολογία 3 του εισηγητήου με την προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία, όχι, ωραία, οπότε την ψηφίζουμε, το, το, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τελική ψηφοφορία άρχεται ε, ε, έναξη της ψηφοφορίας ε, ψηφίσατε πέρα της ψηφοφορίας 35 υπέρ μία αποχή καμία κατά, υιοθετήθηκε συγχαρητήρια κύριε Τζίλε. Τώρα έχουμε προτρέξει του χρόνου και, και ξέρω ότι τα μέλη μας μπερδεύονται όταν ε, ολοκληρώνουμε την εργασία μας νωρίτερα από ό,τι έχει προβλεφθεί. Αυτό πραγματικά είναι ε, παραδειγματικό για την Επιτροπή μας, ε, διότι συνήθως όλοι καθυστερούν, όχι προτρέχουν. Και τώρα είναι η σειρά του κυρίου Φλέκενστάιν για τον κανονισμό, τον οργανισμό ΕΜΣΑ, ασφάλεια στη θάλασσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο για τον κανονισμό της ΕΜΣΑ, του ΕΜΣΑ μάλλον, δεν ήταν εύκολες. Κανένα δεν περίμενε να είναι εύκολες. Οι δύο μεγάλες ε, χώρες δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να συμφωνήσουν ε, στον ε, συμβιβασμό. Η Δανική Προεδρία προσπάθησε έντονα να καταλήξουμε σε συνετές, ε, λογικές ε, διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο σας συστήνω να εγκρίνετε, να υπερψηφίσετε. Θα αναφέρω 7 σημεία τα οποία για μας είναι σημαντικά. Καταρχάς, ο, οργανισμός, ο κανονισμός αυτός θα καλύπτει και ε, τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στις υπερπόντιες πλατφόρμες ε, άντλησης πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομική βάση, αλλά ζητήσαμε από την Κομισιόν να επεξεργαστεί τη νομική βάση για την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων από τις πλατφόρμες και στις πλατφόρμες αυτές για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ακριβώς αυτή τη νομοθετική βάση. Το τρίτο σημείο είναι η αυξημένη συμμετοχή ε, του ΕΜΣΑ στην καταπολέμηση της πειρατείας όπου θα προσφέρει την τεχνική της υποστήριξη. Αυτό δεν είναι τίποτα καινούριο, αλλά κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ε, ήταν κάπως παράδοξο ότι παρόλες τις προσπάσεις που έχουν γίνει υπήρχαν ακόμα προβλήματα στην έγκριση, δηλαδή στη συμφωνία μέσα στο Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει η... το ΕΜΣΑ θα προσφέρει την τεχνική υποστήριξη όπου μπορεί στο θέμα της πειρατείας. Τέταρτο σημείο, ε, νομίζω το είχαμε συζητήσει αυτό και ήταν δική μας επισημία να ασχοληθεί για τη μείωση της ε, διοικητικής γραφειοκρατίας στην αυσιπλοεία. Ε, τώρα το ΕΜΣΔΑ θα μπορέσει να διαθέσει τα στελέχη του, την υποδομή του για να μπορέσουμε να, ενισχύσουμε την ε, ναυσιπλοεία και την αυτιλία την ευρωπαϊκή με μείωση της γραφειοκρατίας. Το επόμενο σημείο είναι βέβαια η το, οι ναυτεργάτες ε, το, και οι ναυτικοί συνθήκες εργασίας ε, ε, κλπ. όπου θα μπορεί να συντονίζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση των εργαζομένων αλλά ό,τι υποστήριξη θα παράσχει το έμψα σε αυτό το τομέα θα γίνεται ε, εθελοντικά, όχι υποχρεωτικά. Θα είναι εθελοντική συμμετοχή. Επίσης συζητήσαμε κάτι το οποίο για μένα ήταν προφανές, αλλά για τους άλλους δεν ήταν, ότι η πολιετής στρατηγική του ΕΜΖΑ θα πρέπει να συζητηθεί εδώ, σε μας. Εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή. Έτσι καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική πρόταση. Ευχαρίστησα στον ομόλογό μου από τη Δανική Προεδρία, από τους εκπροσώπους της Κομισιόν και από το σκιώδη, τους σκιώδης εισηγητές, οι οποίοι συνέβαλαν στο να διευκολύνουν το έργο μου. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο κύριος Σιγάντης από το ΕΛΚ, παρακαλώ τώρα, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αρχίζω με τον είμαι δίκαιο. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Και δεν το λέω επειδή ήθιστε, το λέω γιατί πραγματικά το πιστεύω. Και αυτός είναι και ένας ε, από του κύριους λόγους που έχουμε επιτυχία. Η ελαστικότητα δηλαδή. Και πιστεύω ότι δείχνοντας ελαστικότητα εισηγητής καταλήξαμε σε αυτή την επιτυχία. Πρέπει όντω να είμαι δίκαιο επίσης και απέναντι στην Επιτροπή. Να πω ότι και αυτή ήταν ε, ευέλικτη και βοήθησε να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε εδώ διάφορες πτυχές όσον αφορά την συγχρηματοδότηση αυτή που έχουν τη σημασία τους. Πρέπει να υπογραμμίσουμε πρώτα απ' όλα τη συνεργασία με διαφορούς εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη επιτυχία για μας, για την Ευρώπη δηλαδή. Δεύτερον, υπάρχει βελτίωση στην κατάρτιση των αυτεργατών για να αποφεύγονται ατυχήματα και για να υπάρχουν καλύτερες επιδόσεις στις θαλάσσιες μεταφορές μας. Επίσης, βοηθήσαμε να φτιαχτεί ένας ευρωπαϊκός ε, θαλάσσιος χώρος χωρίς σύνορα, κάτι το οποίο ενισχύει δίχως άλλος τη λειτουργία του τομέα. Η ΕΜΣΑ πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει επίσης και για την μείωση απορρίπανση στην περίπτωση τέτοιων ε, πλατφόρμων εξόριξης με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις στα νυχτά της θάλασσας εφόσον θα έχει νέες δραστηριότητες και αρμοδιότητες στα θέματα ασφάλειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμφωνηθεί και πιστεύω ότι η επιτυχία που έχουμε μέχρι τώρα οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στον εισηγητή, ο οποίος εκφράζει το κοινό αίσθημα. Δεν ήταν εύκολο, γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι ο εισηγητής έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά πέτυχε και πρέπει όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι. Η δικιά μου πολιτική ομάδα πάντως είναι από το αποτέλεσμα αυτής της διαλλαγής. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Κυρία Μπίλτα, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για την ηρεμία του, για τον τρόπο ε, που διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, έγιναν πολλές προσπάθειες για να εμείνει στη θέση του απέναντι σε διάφορα μέλη του Συμβουλίου. Με το σχέδιο αυτό ενισχύονται οι αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ. Είναι αυτός ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε και να κοιτάξουμε το μέλλον προλαμβάνοντας νέες καταστροφές. Πιστεύω ότι Πιστεύω λοιπόν ότι στο θέμα της καταπολέμησης της ρήπανση, όταν μιλάμε για τις πλατφόρμες εξόριξης πετρελαίου πρέπει να μείνουμε στην πρότασή μας. Η ομάδα μας θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι κατάλληλες εγγύησεις και η νομική βάση έτσι ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον ρήπανση από τέτοιες πλατφόρμες. Όσον αφορά την κατάρτιση, εδώ η κατάρτιση και η συνεργασία αναφέρεται σε θελοντική βάση δυστυχώς για μας. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται εναρμόνιση στην κατάρτιση των αυτεργατών. Και εμείς θα θέλαμε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή σχολή κύρους που να δείχνει και ότι η Ευρώπη έχει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των, ε, της ρήπανσης για παράδειγμα. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Ελπίζω στο μέλλον να τα καταφέρουμε. Θα θέλαμε δηλαδή να δεσμευόντουσαν ε, τα κράτη-μέλη στο θέμα της εναρμόνισης της κατάρτισης των ναυτικών. Τέλος, υπάρχει και μια πτυχή την οποία εμείς επικρίναμε στις διαπραγματεύσεις. Ε, θα σας πω περί την πρόκειται. Είναι η πρόταση του Συμβουλίου που έλεγε ότι αν υπάρχει συμφωνία στο γενικό πακέτο θα ήταν διατεθειμένοι να συμπεριλάβουν τις τροπολογίες ή τους συμβιβασμούς τέλο πάντων που έχουν να κάνουν με την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να μπαίνουν προϋποθέσεις στο να συμπεριληφθούν τροπολογίες ή συμβιβασμοί για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή είναι μια παράμετρος που δεν έχει μπει στις διαπραγματεύσεις ποτέ μέχρι τώρα εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι δηλαδή μια αντίφαση για μένα όταν ε, ακούμε την Επίτροπο Ρέντινγκ να προσπαθεί να πιέσει το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τον ίδιο αριθμό αντρών και γυναικών. Αυτή είναι η κριτική που έχω να κάνω. Θα θέλαμε να είχαν συμπεριληφθεί περισσότερες τροπολογίες. Εκεί, για παράδειγμα, που λέω ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσουν να έχουν ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς θα θέλαμε να είχαμε πάει ακόμα πιο πέρα. Για να υπάρχει συνέπεια με τις πολιτικές, τις ευρωπαϊκές και της Επιτροπής και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την ισότητα. Τέλος πάντων, γενικά μιλώντας πάντως, εκτιμώ θετικά το αποτέλεσμα, γιατί παρόλα αυτά καταφέραμε να φτάσουμε πιο μακριά από ό,τι φανταζόμασταν στην αρχή και είμαστε πεπισμένοι ότι η πραγματικότητα θα μας υποχρεώσει να ε, αντιμετωπίσουμε καλύτερα και να προσαρμόσουμε ακόμα καλύτερα τις προδιαγραφές της ΕΜΣΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, μια που ευχαριστούμε, ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Φακεστάιν για την τόσο επικοδομητική του στάση, για την έκθεσή του και για το ότι στήριξε τον δικό μας ενθουσιασμό για τις αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ προκειμένου να ασχοληθεί και με τις πλατφόρμες εξόριξης πετρελαίου. Είναι πολύ θετικό αυτό για το μέλλον. 100% συμφωνώ για αυτά που είπε η προλαλή σας όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μα μετά τη Λισαβόνα θα πρέπει τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Δεν είναι όμως. Είναι ευαίσθητο το θέμα, αλλά πράγματι ούτε καν μιλάνε πολλές γυναίκες για τις πλατφόρμες. Είναι μια χαμένη ευκαιρία, νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία και σε αυτό το θέμα. Αυτά. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Φαλκενστάιν. Ευχαριστούμε. Ναι, ε, άλλος για να επιβεβαιωθεί το θέμα των δύο φίλων. Α, εσείς. Κύριο Ζήλε. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του κύριου Φαντάλεν, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Φακεστάν για τις προσπάθειες που έκανε μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες δηλαδή της ΕΜΣΑ, οι οποίες ενισχύονται και όσον αφορά επίσης και το θέμα της καταπολέμησης της ρήπανσης από τις πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και γενικότερα για τις προσπάθειες που γίνονται όσον αφορά το θαλάσσιο χώρο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φακεστάν και εγώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τούσας δεν είναι εδώ. Άρα εδώ τελειώνει ο κατάλογος των ομιλητών. Εκτός αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Ο κύριος παρακαλώ. Ε, δεν χάνετε ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ εκ μέρους της ομάδας μου θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Εισηγητής για ολόκληρο το κοινοβούλιο βέβαια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειες που έκανε και για το συμβασμό στον οποίο κατέληξε. Η ομάδα μου θέλει επίσης να υπάρξουν εξελίξεις στο θαλάσσιο χώρο, ένα θαλάσσιο χώρο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αυτή πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή περισσότερο κοινή διαχείριση του θαλάσσιου χώρου και πιο συντονισμένος ε, ρόλος για να αντιμετωπιστεί η πειρατεία. Όντως, ο ρόλος που αναλαμβάνει η ΕΜΣΑ για την καταπολέμηση της ρήπανσης είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να πάμε ακόμα πιο πέρα. Οι εθνικές αρχές πρέπει επίσης να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες αρμοδιότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Και εγώ συγχαίρω τον εισηγητή. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γέγκερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκ μέρου του κύριου Καραμίτσου, τον οποίο καθιστώ σήμερα εδώ, Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μας για την Συμφωνία Δεύτερης Ανάγνωσης. Πρώτα απ' όλα, χαρητήρια και από μένα στον εισηγητή, τον κύριο Φλακενστάιν, και στους συνεισηγητές για τον τρόπο, τον τόσο επαγγελματικό με τον οποίο αντιμετώπισαν αυτό το θέμα. Γι' αυτό και στηρίζουμε απόλυτα το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ένας λογικός και καλός συμβιβασμός, όπως ακούσαμε και πριν. Η Επιτροπή ε, Πάντα, όπω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλει μια πιο φιλόδοξη απόφαση. Ο συμβασμό όμω καλύπτει ε, τα κύρια στοιχεία τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εντολή, δηλαδή, η οποία επιτρέπει στην ΕΜΣΑ επιτυχώ να συνεισφέρει και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Αναλαμβάνει νέα καθήκοντα και θα συνεχίσει να ασχολείται με τις θαλάσσιες μεταφορές χωρίς σύνορα, την καταπολέμηση της πειρατείας και θα παίξει και έναν ρόλο όσον αφορά τα ferry boats. Θέλουμε επίσης, θέλαμε μάλλον επίσης να δώσουμε και μια απάντηση στο θέμα της ρήπανση από τις πλατφόρμες εξόρυξης κλπ. Δεν μπορέσαμε δυστυχώς να πείσουμε το Συμβούλιο να επεκτείνει περισσότερο τις αρμοδιότητες αυτές και ε, offshore, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται όσο προχωράμε και έχουμε την έκθεση πρόοδου να ασχοληθεί με αυτό παρετέρω. Είναι πολύ καλό λοιπόν το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να δούμε περισσότερο τι θα κάνουμε με τις εγκαταστάσεις offshore. Εμείς επίσης πρέπει να σας πω ότι στηρίζουμε τη διατύπωση για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια που είπατε για τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τελικό συμβιβασμό και προσδοκούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής, κύριε Φράγκεσταν, έχετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συνεργασία. Αυτό και μόνο. Καλώς. Θα γράψω στο Συμβούλιο, εκφράζοντας την ε, συμφωνία μας. Αυτοί θα επανέλθουν και μετά θα ψηφίσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Φλέκεντσαν. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ακρόαση που έχουμε για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη 10 και μισή με την Ήτρα. Στην άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να πάμε. Στην αίθουσα 3C050. 10 και μισή να είσαστε εκεί. Καλύτερα θα ήταν να μην πάμε εμείς οι τρεις, ε, να είσαστε όλοι στην ακρόαση αυτή. Δέκα και μισή λοιπόν. Επίσης, υπενθυμίζω ότι στις 3 πρέπει να έρθουμε εδώ. Για να μιλήσουμε με τον κύριο Γιαζεμπόφσκι. Κυρία Γιάλα Σέντερ, κάτι θέλετε να πείτε. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να πω οι συνάδελφοι να έρθουν στην ακρόαση αυτή. είναι πολύ σημαντικό γιατί θα συζητηθούν τα παραρτήματα και μόνο αν οι ευρωβουλευτές έρθουν και είναι παρόντες και μα πούνε τις προτάσεις τους θα τι λάβουμε υπόψη μας. Τέλο πάντων, σαν προειδοποίηση το λέω, να ξέρετε ότι αν δεν είσαστε εκεί ε, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε υπόψη μας και τα όσα θα προτείνετε. Ωραία, ξεκάθαρο αυτό. 10 και μισή θα λέμε εκεί λοιπόν.